Πρόεδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Από πλευράς της ε, Αντιπροέδρου της ε, Επιτροπής ε, θα λάβει τον λόγο ο εκπρόσωπος. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο ε, για αυτή την πολύ σημαντική και επίκαιρη συζήτηση ώστε να συζητήσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Θα πρέπει να το πούμε ότι η Ιεμένη έχει παραμεληθεί, ε, πρόκειται για μια ξεχασμένη κρίση και είναι απαραίτητο να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό που έχει περιγραφεί ως μια ανθρωπιστική κρίση καταστροφικών ε, ε, καταστροφικής κλίμακας όπου ο κόσμος χρειάζεται άμεσα βοήθεια. Παρά την επανειλημμένη διεθνή καταδίκη, πιστώνουμε ότι συνεχίζονται να συνεχίζεται η παραμέληση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πολίτες και η άμαχος πληθυσμός γίνεται στόχος από όλες τις πλευρές της σύραξης σχεδόν καθημερινά. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις πρόσφατες ε, επιθέσεις κατά των γιατρών χωρίς σύνορα και των εγκαταστάσεών τους στην Ιεμένη που δέχτηκαν επιθέσεις και υπέστησαν ε, θύματα. Ακόμα ένα παράδειγμα της παραβίασης της διεθνούς νομοθεσίας που γίνεται στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Η ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης διαρκώς αυξάνεται. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι 21,2 εκατομμύρια Ιεμενίτες ε, ε, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τη στιγμή 14,4 εκατομμύρια υποφέρουν από υποσυτισμό και 9,3 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και ε, υγειονομική περίθαλψη. Θα πρέπει να αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους ε, Ιεμενίδες και αυτό προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Στο ανθρωπιστικό μέτωπο η Κομισιόν ε, αύξησε κατά 17 εκατομμύρια ευρώ το βοήθεια προς τη χώρα, φέρνοντας έτσι το ποσό στα 52 εκατομμύρια ευρώ για το 2015. Ορισμένα κάτι μέλη ήδη συμβάλλουν με βοήθεια ανθρωπιστική και επίγουσα βοήθεια και περισσότεροι θα αυτό εφαλεί τα πιο ευάλωτα άτομα, τους εσωτερικά εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες που έχουν ε, ε, ε, εγκλωβιστεί στην Ιεμένη και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική και την επιστηστική κρίση, των οποίων η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της σύραξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα μέρη ώστε να επιτρέψουν την πρόσβαση για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, το επίπεδο της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης είναι μόνο η μια πτυχή, Αυτό το γνωρίζουμε γιατί ο πληθυσμός εξαρτάται από τις εχογές για το 90% της κάλυψης των βασικών αναγκών και η άρση των εμπορικών ε, ε, περιορισμών είναι εξίσου σημαντική. Ε, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕ αλλά και τους άλλους εταίρους ώστε να επιταχύνουμε τους μηχανισμούς ε, εποπτείας και επιθεώρησης ώστε να επιτραπεί η ροή ανθρωπιστικών και εμπορικών αγαθών στο οποίο συμβάλλουμε με 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο δρόμος είναι ο πολιτικός δρόμος, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο δεύτερο ήμιση του 2014 και κυρίως μετά από το Μάρτιο του 2015 έχουν σοβαρά βλάψει τις επιτυχίες αλλά και την εφαρμογή της ε, μετάβασης της και έχουν αφήσει τη χώρα στο χείλος της ανθρωπιστικής καταστροφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε στα συμπεράσματα του Σεπτεμβρίου 2015 ότι πιστεύει πως οι λύση σε αυτή την κρίση θα πρέπει να είναι πολιτικής φύσης ε, καθώς και μια πολιτική ρύθμιση που θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πρωτοβουλία της GCC, το, αποτέλεσμα του διεθνούς διάσκεψης αλλά και του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας που είναι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί η κατάσταση του λαού της Ιεμένης. Μετά από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στη Γενέβη τον Ιούνιο, έγιναν και ε, ε, ένας δεύτερος γύρος στην Ελβετία ε, πιο πρόσφατα και εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε πλήρως το ρόλο μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει άλλη μια διαπραγμάτευση τις επόμενες μέρες. Στη σύραξη τώρα συμμετέχουν διάφοροι περιφερειακοί ε, παράγοντες και θα ρίνουμε όλους τους παράγοντες αυτούς να παίξουν ε, θετικό ρόλο για μια διαρκή και μόνιμη πολιτική φύση σε λύση. Ε, εμείς ανησυχούμε για την εφαρμογή άμεσων βημάτων ώστε να ε, ισχύσει πάυση πυρός, ε, που πράγμα που επιτεύθηκε και παλιότερα, αλλά παραβιάστηκε από διάφορα μέρη, ενώ θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή, ε, σεβαστός μάλλον ο νόμος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρξει πρόσβαση κυρίως στην πόλη Ταΐσε αλλά και στη Σάντα και όλες τις άλλες περιοχές που έχουν πληγεί. Ε, στην Ιεμένη η κατάσταση είναι δραματική. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη λογοδοσία για όλες τις ε, βιοπραγίες. Ε, ε, το Συμβουλίο Ασφαλείας υιοθέτησε ένα συμβαστικό ψήφισμα τον Οκτώβριο 2015 για τεχνική βοήθεια και δημιουργία δυνατοτήτων για την Ιεμένη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεσπίζει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας Εθνικής Επιτροπής Έρευνας που αναμένει ο ΙΕ να εργαστεί ανεξάρτητα. Εγώ επαναλαμβάνω τη δική μας έκκληση για ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των ε, παραβιάσεων της Διεθνούς Νομοθεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Περιμένουμε πλήρη ενημέρωση στην 31η Σύνοδο του Συμβουλίου και μια συνολική γραπτή έκθεση στην 23η Σύνοδο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Και περνάμε τώρα στους αγορητές ε, για τις ομάδες. Ε, η πρώτη θα είναι η κυρία Μαρία Γκάμπριελ. Ένα μισή λεπτό <clears throat> για το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφοι, έχουμε τριπλή επίγουσα κατάσταση. Είναι πολιτική ανάγκη, ασφαλική και ανθρωπιστική. Η κατάσταση ανθρωπιστική λόγω των συγκρούσεων είναι χειρότερη από ό,τι στη Συρία μετά πέντε χρόνια. Είναι από τι κρίσει ανθρωπιστικέ σοβαρότερε τώρα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η πολιτική δέσμευση και η προσπάθεια δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την κατάσταση την πραγματική. Θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα να συμβάλλουν περισσότερο στον αθωρημένο σχέδιο τη βοήθεια ανθρωπιστική. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά η ανθρωπιστική βοήθεια, να είναι αμερόληπτη όσον αφορά του πολίτε που είναι του αμάχου που είναι θύματα του εμφυλίου πολέμου. Ε, υπάρχει διπλή απειλή όσον αφορά την ασφάλεια. Έχει χρεκοπήσει το κράτο και ο φίλο πόλεμο ε, είναι κάτι που χρησιμοποιεί τον Ντάεσ και η Αλκάιντα. Και υπάρχει πραγματικό κινδύνο, όπω ανέφερα, που είναι η επέκταση ε, και συμμετοχή κι άλλων φορέων ασταθεία. Η Εμένη συνδέει την Αραβική Χερσόνησο με την Αφρική. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να προβλέψουμε και ποιε κίνδυνε δημιουργούνται. Ε, λοιπόν, όσον αφορά το πολιτικό σχέδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να παίξει σημαντικό. Δύο παρατηρήσει. Από τη μία πλευρά θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τι προσπάθειε του ΟΗΕ, ώστε διαπραγματεύσει να ξεκινήσουν και να κάνουμε περισσότερο ώστε η Εμένη να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη συζητήσεων. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά μεσομεχροπρόθεσμη άποψη, να επενδύσουμε περισσότερα όσον αφορά την ενίσχυση των σχέσεών μα των πολιτικών με τι χώρε του κόλπου και τι ε, του Αραβικού Συνδέσμου για να δημιουργήσουμε συνεργασία. Χωρί αυτά ε, θα δείξει ότι δεν έχουμε λάβει μαθήματα από τι συγκρούσει ε, που έχουν συμβεί σε χώρε τη ε, Αραβική Άνοιξη. Και υπάρχει, έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία να ακολουθήσουμε σωστή προσέγγιση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο είναι ο κύριο Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ για δύο λεπτά εξ ονόματο των Σοσιαλδημοκρατών. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν μια ανθρωπιστική κρίση προέρχεται από μια σύραξη, πολεμική, ιδιαίτερα όταν είναι εσωτερική αυτή η σύραξη σε μια χώρα, ένας εμφύλιος πόλεμος, ο κύριος στόχος πρέπει να είναι να πάψουν οι εχθροπραξίες και να μπορέσει να επιτευχθεί η ειρήνη δίκαια και διαρκέστερη. Διότι βλέπουμε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι πρώτον η απώλεια ανθρώπινων ζώων σε μια τέτοια κατάσταση, δεύτερον η, η καταστροφή θεμελιωδών υποδομών που αφορούν τις ίδιες τις ανάγκες εκείνων που έχουν δυνα... μικρότερες δυνατότητες πρόσβασης στο πόσιμο είδο νερό στην εκπαίδευση και στις υγειονομικές ε, υπηρεσίες και η απώλεια ευκαιριών για μια ολόκληρη γενεά. Τέλος. Και υπό ανθρωπιστικό πρίσμα η διαρκής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η άγνοια των αρχών της αρχής, περιφρόνηση των αρχών της ανθρωπιστικής δράσης και όλα αυτά συμπυκνώνονται σε μια κρίση, στην κατάσταση δηλαδή που ζούμε και βιώνουμε στην Ιεμένη. Όπως επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου και πάλι σε αυτή την περίπτωση και σε σχέση με την Επιτροπή στην Ιεμένη υπάρχουν ανάγκες που πραγματικά πλήττουν 80% και πάνω από τον πληθυσμό, πάνω από 20 εκατομμύρια πολιτών. Και υπάρχουν διαρκείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ομάδα μου και ιδιαίτερα εγώ ως υπεύθυνο για την ανθρωπιστική δράση εισηγητής, μόνιμος εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Συμβουλίου τον Απρίλιο, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών στην αναζήτηση ειρήνης, ειρηνικής λύσης, ασφαλούς και διαρκε, δια, μεγαλύτερης διάρκειας και με την δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση για την ανθρωπιστική βοήθεια προς πελασιμότητα ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εκατομμυρίων ανθρώπων που αυτή τη στιγμή στερούνται και τις πιο θεμελιώδεις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια ο κύριος Charles Τένοκ για την ECR. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, μία από τις πιο φτωχές ε, τις χώρες του κόσμου που ε, ε, εξαρτάται από πάνω από 90% με εισαγωγές για τις επιστημιστικές ανάγκες η Εμένη αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική κρίση και στην αξιολόγηση της κατάστασης είναι δίνες οι προοπτικές, ζωφερές οι προοπτικές. Δόθηκαν πολλά χρήματα στην βοήθεια και η δική μου χώρα πάνω από 250 εκατομμύρια λίρες στερλίνες δώσαμε για αυτή την βοήθεια. Τώρα τίθεται το θέμα της ε, χορήγηση βοήθειας μια και υπάρχουν βομβαρδισμοί και καταστρέφονται τα πάντα από τα αεροπλάνα της Σαουδικής Αραβίας ε, και βλέπουμε καταστροφή υποδομών ε, πλήττονται ήδη, ήδη οι άμαχοι από τους Σαουδάραβες γιατί δεν στοχεύουν καλά στου βομβαρδισμούς του στα πολεμικά του αεροπλάνα και έχουμε πάμπολα θύματα υπάρχει αντιμετω... τοπική αντιπαράθεση της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν για την τοπική τοπική επικυριαρχία, περιφερειακή επικυριαρχία και τα δυνάτα υφίστανται άλλοι όπως σε αυτό τον πόλεμο ε, δι' αντιπροσώπων στην Ιεμένη. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια για δύο λεπτά η κυρία Μαρία Τσεσάκε παρακαλώ για την Άλντε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ. Ο λαό στην Ιεμένη πεθαίνει από ασθένειε και από την πείνα και εξαλείφω του βομβαρδισμού από τη συμμαχία τη οποία ηγείται η Σαουδική Αραβία. Ακολουθείται από τη ΣΥΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Πρωθυπουργό Κάμερο αυτή την εβδομάδα είπε ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η δουλειά που κάνει η Σαουδική Αράβια έχει συγκεκριμένο στόχο. Προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν λειτουργεί. Είναι μια ντροπή ότι οι προτάσεις σας, και μιλώ, οι προτάσει τη να γίνει έρευνα για τους ε, εγκλήματα πολέμου στην Ιεμένη που θα εξεχθεί μέσω του ΙΕ και κάτι που το σαμποτάρισε η Σαουδική Αραβία και ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποστήριξαν την Ολλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να είναι ισχυρή, χρειάζεται μια κοινή θέση. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μιλήσατε για την εξαγωγή τη σταθερότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αξιέπαινο στόχο. Θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προσπαθήσει να σταματήσει την εξαγωγή όπλων προ τη Σαουδική Αραβία. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω κατά πόσο είσαστε πρόθυμο να κινηθείτε προ ένα εμπάργκο προ το Συμβούλιο τουλάχιστον βομβών, ε, μαχητικών αεροσκαφών και μαχητικών ελικοπτέρων και κατά πόσο θα ασκήσετε πιέσεις οποιονδήποτε ίσως να χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς οι οποίες είναι δυσανάλογο ε, όπλο και χρησιμοποιείται σύμφωνα σχετισμού στην Ιεμένη. Συμφωνείτε ότι η βία στην Ιεμένη δείχνει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει τη σχέση τη με τη Σαουδική Αραβία και να είναι πιο ισότιμη η αντιμετώπιση ε, σε σχέση με που έχουμε με το Ιράν. Μετά τη συμφωνία για τα πυρηνικά υπάρχει περιθώριο να συνομιλήσουμε αυτή τη χώρα με το Ιράν δηλαδή για να σταματήσει και η βία στο, στην Ιεμένη. Το Ιράν όπως και η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να προωθηθούν για να συμμετάσχουν στη λύση και να σταματήσουν οι βιοπραγίες στη Μέση Ανατολή. Τέλος, ε, ε, οι αποκλεισμοί, οι θαλάσσιοι και οι αέρια έχουν παρεμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια να χορηγηθεί και είναι κάτι που χρειάζεται και αυτό σκοτώνει ανθρώπους, συμφωνώ με τους γιατούς χωρίς σύνορα. Διατείνονται ότι σταματήσαν να έρχονται οι άνθρωποι στα νοσοκομεία διότι πιστεύουν ότι τα νοσοκομεία αποτελούν στόχους και φαίνεται να είναι ανησυχητικό φαινόμενο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ <clears throat> κυρία Σάρτια. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Τενόκ. Την δέχεστε. Μάλιστα, εντάξει, κύριε Τένο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πλεκάτα. Αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο υποθέτω για την αρνησή κυρία όσον αφορά τις εξεταστικές δράσεις που προτάθηκαν από την ε, Ολλανδία για εγκλήματα πολέμου στην Ιεμένη. Έχετε κάποια τεκμήρια για το ότι εσκεμένα ε, σκόπευσαν ε, οι Σαουδάραβες άμαχους. Αν έχετε τέτοια τεκμήρια γιατί δεν τα δημοσιεύετε. Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία και υπάρχει πραγματικά ισχύνη να πιστέψει κανείς ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύει κάποιους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε και για την ερώτησή σα. Δύο παρατηρήσει υπάρχουν στη όσα είπα που ίσω οδήγησαν σε κάποια παρανόηση. Πρώτον, από την Ολλανδική κυβέρνηση και από πλευρά του κ. Κούρνες μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό, υπήρξε η εκτελεστική εντολή των Ηνωμένων Εθνών που είχε τροχοπεδηθεί και θα έλεγα δυστυχώ διότι εδώ η εξέταση για αυτά τα εγκλήματα έχει σημασία κλειδιού πραγματικά. Και τώρα για το τι συνέβη με τα νοσοκομεία είναι κάτι το οποίο οι αρμόδιοι ε, μη κυβερνητικέ ε, ε, υπηρεσίες, μη κυβερνητικέ οργανώσεις των ιατρών χωρίς σύνορα τις έκαναν. Έτσι λοιπόν εδώ σε αυτό υπάρχει αναφορά για αυτό το οποίο συνέβη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Υπάρχει δεύτερη μπλε κάρτα. Σας προτείνω ωστόσο <clears throat> για αυτό το χρόνο να λάβουμε μόνο μία μπλε κάρτα στην παρέμβαση και γι' αυτό λοιπόν κάποια άλλη φορά θα παρέμβετε εσείς με την μπλε κάρτα σας. Επόμενος αγορητής η κυρία Φερζιά. <coughs> για την ε, ομάδα UGL. Παρακαλώ ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2011 είχε λεκά κινήματα το 2011, αλλά μετά από αυτό έχει μπλέξει σε θανατηφόρο σύγκρουση εμένη και κινητοποιούνται, έχουμε τη μία ε, τη Σαουδική Αραβία και από την άλλη τις δυνάμεις του Προέδρου Σαλέ. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το δίπολο αν θέλετε. Και θέλω να ότι είναι μόνο εσωτερική σύγκρουση μεταξύ των Σιτών και των Σουνιτών. Ε, οι Σουνίτες στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, άλλοι από το Ιράν. Αγνοούμε έτσι την ιστορία της πόλης, οι συμμαχίες που υπάρχουν, ότι είναι περίπλοκη η πολιτική κατάσταση και κοινωνική εκεί. Και είναι ασφαλές. Ο πληθυσμός της Ιεμένης είναι από τους στον κόσμο. Βρίσκεται σε υποανάπτυξη, βρίσκεται ανάμεσα στις συγκρούσεις των δύο πλευρών. Και τελικά είναι πολύ επιθετική η Σαουδική Αραβία με μεσονικέ αντιλήψει. Και εμεί εθελοτυφλούμε μπροστά τα συμπεριφορά τη Σαουδική Αραβία. Μέχρι, πότε θα λησμονούμε την Ιεμένη. Θα πρέπει να διορθώσουμε τα σφάλματα που κάναμε τη Συρία. Δεν θα πρέπει να αρκούμε σερβιστική βοήθεια σε καταγγελίε, να δράσουμε έναντι εκείνων που διαπράττουν τι πράξει, να μην κρυβόμαστε πίσω από τον ε, ΟΗΕ. Σα ευχαριστούμε κυρία Βρέζα. Από τους Πρασίνους στη συνέχεια η κυρία Μπάρμπαρα Λοκμπίντερ παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από το Μάρτιο 2015 κλιμακώνεται η σύραξη στην Ιεμένη και έχει περιπέσει σε μια ανθρωπιστική καταστροφική κατάσταση η χώρα. Οι άμαχοι είναι εκείνοι που υποφέρουν. Πάνω από δύο εκατομμύρια παιδιά που υποσυτίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν άμεσα ώστε επαρκή επισητιστική βοήθεια να εξασφαλιστεί για την Ιεμένη. Στην σύραξη της Ιεμένης έχουμε δύο ευάλωτε συμμαχίε Στο βορρά οι επαναστάτες που συνδέονται συνδέονται με τον πρώην πρόεδρο Σάλι και έχουμε και την ε, προσπάθεια των ε, αποσχιστικών δυνάμεων στο Νότο. Όσο και πιο περίπλοκη είναι η σύραξη αυτή, ε, δημιουργείται ακόμα μια περιπλοκή επιπλέον με την ανάμειξη Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Υπάρχει άμεση εμπλοκή με την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας που πλήττει στόχους. Έχουμε χιλιάδες αμάχους που έγιναν θύματα αυτών των επιθέσεων επιθέσεων καθώς επίσης και από τους επαναστάτες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άμαχοι ως στόχοι, νοσοκομεία, αποθήκες. Εδώ πραγματικά απαγορεύεται και η χρήση των βομβών ε, διασποράς και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε και εμπλοκή και του Νταέσ και του ΙΚΙΣ Ισλαμικού κράτους Ιράκ και Συρία ζητούμε από τους εμπλεκόμενους να πάψουν αυτές τις εχθροπραξίες αντί περαιτέρω κλιμάκωσης ε, της βίας ε, και παροχής όπλων ε, πρέπει να αναζητηθεί πολιτική λύση μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, για δύο λεπτά, ο κύριος Καστάλντο στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποσιωπήσουμε την εσωτερική διχόνοια. Συχνά είναι το να εστιάσουμε την προσοχή στον εξωτερικό εχθρό, απέναντι στον οποίο κάθε άλλη απόκληση θα πρέπει να αφαιθεί κατά μέρο. Ε, μπορεί αυτοί να θεωρηθούν προδότες ή τρομοκράτες όσοι δεν υποκύπτουν σε όλα αυτά. Ε, η χορηγή της μειονότητας ούτε στην Ιεμένη είναι το Ιράν. Όμως δεν πάνε τα πράγματα όπως είχαν προγραμματιστεί. Ε, η κατακτήση του Άντεν και του Τουπά που είναι κρίσιμα για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ Χελμαντάντ οδήγησαν σε χιλιάδες νεκρούς, το 60% λόγω των αδιάκριτων αεροπορικών επιδρομών, 3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, 16 εκατομμύρια Εμενητών χωρίς ε, νερό και εντωμεταξύ το κράτος ε, πτωχεύει. Ε, αυτό που είναι ακόμα πιο σοβαρό είναι ο πολύ ψηλός αριθμός παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επαληθευτεί από τον ίδιο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών όταν ήδη η συμμαχία ήταν υπό την αιγίδα του ψηφίσματος του ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας Μπανκιμούν αρχίζει να εκφράζει αμφιβολίες για την διαχείριση της Σαουδικής Αραβίας. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή πριν να ξεκινήσει μια επίσημη έρευνα. Το μήνυμα που πρέπει να γίνει είναι αυτό. Δεν θα ήθελα να σκέφτομαι ότι όλες αυτές, ε, όλη, αυτή, όλη αυτή η αφηρημάδα των Ευρωπαϊκών κρατών και των Ηνωμένων Πολιτειών που πολύ συχνά ε, ε κάνουν ε, τα στραβά μάτια είναι το τίμημα για να, που θα πρέπει να πληρώσουν ε, σε σχέση με ε, την πυρηνική δύναμη του Ιράν. Θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια για μια ειρηνευτική διαδικασία και να ακολουθηθεί πολύ αυστηρή γραμμή στο να καταδικαστούν οι βιοπραγείς και στο να ζητηθεί έρευνα. Γιατί κλείνοντα τα μάτια για να προστατεύσουμε αυτό που μας είναι χρήσιμο θα φαίνεται σαν να έχουμε τυφλωθεί απέναντι στο απολύτως απαραίτητο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι τώρα ο κύριος Νικόλα Μπέι για ένα λεπτό. Στη δήλωση της 10ης Δεκεμβρίου η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, καταδίκασε τη νέα, τον νέο βαδρασμό ενός νοσοκομείου στα βόρεια της Ιεμένης που προκάλεσε έξι νεκρούς και πολλούς σοβαρά τραυματισμένους μεταξύ των οποίων και μέλη των γιατρών χωρίς σύνορα. Μίλησε για επιθέσεις που ηθελημένα στοχεύουν ανθρωπιστικές ε, επιχειρήσεις και τους, ε, τον άμαχο πληθυσμό. Όμως δεν ζητάτε την έναρξη έρευνα. Θυμίζω ότι είναι το τρίτο νοσοκομείο το οποίο διευθύνουν οι γιατροί Χωρί σύνορα και το οποίο στοχεύει η Σαουδική Αραβία μέσω της συμμαχίας κατά των Σιητών. Επίσης, δεν σας ακούω να καταδικάζετε τη χρήση των όπλων που και ε, των πυρομαχικών των Σαουδαράβων που απαγορεύονται από τη σύμβαση του ΙΕ. Α, και ξέχασα ότι οι φίλοι μας οι Σαουδάραβες έχουν την Προεδρία του Συμβουλίου ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Αυτή την αγόρασαν με τα πετροδολάρια τους. Ε, η Εμένη ήταν ήδη ένας μεγάλος πολιτισμός, αυτός της ε, βασίλισσας του Σαμπά, για την οποία μιλά και η Παλαιά Διαθήκη. Θα, θα σταματήσουμε να θανατώνουμε τους Ιεμενίτες ε, ή όχι. Αλέσια Μαρία Μόσκα, τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σοβαρότητα τη κατάσταση στην Ιεμένη έπρεπε να επιβάλλει την καλύτερη, πιο στενή συνεργασία μεταξύ των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των διαφόρων εμπλεκομένων μερών και εδώ εκφράζουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανησυχία. Διότι στο, στην πλήρη ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τον πληθυσμό είδαμε ότι να υπάρχουν αντιθέσει μεταξύ εκείνων ε, που θα έπρεπε να είναι στο ίδιο μέρο για να μπορέσουν να βρουν λύσει. Ανησυχούμε κυρίω για αυτό που ζούει ο πληθυσμό στα νοσοκομεία όπω υπενθυμίστηκε ε, λείπουν βασικά φάρμακα και το πρόγραμμα το Παγκόσμιο Διατροφής είδε ότι περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από την πείνα, 6 εκατομμύρια σε απελπισμένη ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι ειδήσει που μαζέψαμε και είδαμε ότι η συμμαχία της οποίας ηγείται Δική Αραβία έχει δημιουργήσει πάλι από 2.500 θύματα αμάχων και έχει επίσης και ε, πλήξει με βομβαρδισμούς και αποθήκες φαρμάκων και απευθύνω μια έκκληση ούτως ώστε να γίνει αμέσω διπλωματική δράση, ούτως ώστε να υποστηριχθεί ο πληθυσμό τη Ιεμένης και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας διάδρομος ανθρωπιστικός με την επιβολή πάψο ε, του πυρός και να δώσουμε νέα όθηση στι ειρηνευτικέ διαδικασίε. Ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σύγκρουση στην Ιεμένη είναι ιστορική. Ε, έχει είναι ιστορική κρίση. Ήμουν εκεί σαν ανταποκριτή πολεμικό στη δεκαετία του 70 και δεν άλλαξε τίποτα. Είναι οι Σιήτες κατά των Σουνιτών, ε, οι ε, με, με τους Χούτις, έχουμε τη Σαουδική Αραβία που παρεμβαίνει ε, κάτι που έκανε από τη δεκαετία του 20 σε διαδοχικές συγκρούσεις. Και υπάρχει μια ιστορική σύγκρουση, μία από τις πολλές που σημειώνται στην περιοχή. Το βασικό πρόβλημα είναι η ομή εγκληματική παρέμβαση Σαουδική Αραβίας. Είναι μια εσωτερική σύγκρουση, ξεκίνησε εσωτερική σύγκρουση που γίνεται σφαγή, γιατί υπάρχουν ηγεμονικοί στόχοι της Σαουδική Αραβίας στην ε, περιοχή. Ε, προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της με χρήση μισθοφόρων. Ε, οι ούτως αποκαλούμενοι ε, είναι υποτίθεται φίλοι μας. Πρέπει να τους πούμε αρκετά. Δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Ιεμένη αν δεν καταφέρουμε να διώξουμε τους ξένους μαχητές από την εμφύλη αυτή σύραξη. Συμφωνώ απολύτως για τη διάσκεψη της ειρήνης. Για να φτάσουμε στη διάσκεψη της ειρήνης θα πρέπει οι Σαουδάραβες που είναι εκεί επιτιθέμενοι να απομακρυνθούν. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος James Χάρμπορ έχει το λόγο. Εγώ είμαι σε στενή επαφή με όλους εκείνους ε, οι οποίοι ε, αναζητούν την ανεξαρτησία στην Νότια Εμένη και παρά τις ε, προσπάθειες δυστυχώς δεν μπορούσαν να καταφέρουν τίποτα έχουν αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν τους Ιρανούς και πολλούς άλλους υποστηριχτές τους κατόρθωσαν να απελευθερώσουν, να του απελευθερώσουν, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται και βλέπουμε ότι οι ακραίες δυνάμεις επανενώνονται. Το κίνημα αυτό κατόρθωσε ήδη να ελέγχει την κατάσταση και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ιεμένη. Ε, Πάντως στην Ιμένη υπάρχουν διάφορες ε, ομάδες, φυλές, ε, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν τάξη, αλλά δεν το επιτρέπει η Σαουδική Αραβία. Ο πληθυσμός υποφέρει διότι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν εξακολουθούν να παίζουν τις δικές τους πολιτικές εις βάρος ε, της Ιεμένης. Κυρία Πρόεδρε, εάν λοιπόν θέλουμε πραγματικά την σταθερότητα στην Ιεμένη, οι διεθνείς παίκτες θα πρέπει να εμπλακούν αντί να περιμένουν τους ε, συνήθεις υπόπτους ε, να δραστηριοποιηθούν σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάρβερ. Ίγκεν Φρόντ για ένα λεπτό. Ενάμιση λεπτό λέει ο κύριος Φρόντ. Όχι ένα λεπτό γράφει εδώ. Συγγνώμη. Ο κύριος Κάρβερ είχε 1,5 λεπτό. Ένα λεπτό εσείς τόσος πόνος κυρία Πρόεδρε και καμία προσπάθεια να μειωθεί. Πρόκειται όμως για μια στρατηγική σημασία περιοχή. 6.000 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί. Και κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι. 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από πείνα. Δεν υπάρχει καθαρό νερό, ούτε ρεύμα. Αυτή είναι η εμένη του σήμερα. Οπότε είναι κατεπήγον να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσεις ταυτόχρονα, πρέπει να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι το ότι οι ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις ε, που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα πρέπει να μπορούν να δουλέψουν ανεμπόδιστα. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υποστηρίξουμε τον ΟΗΕ για να υπάρξει μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μετά ειρήνη, αλλά δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα να εξάγουμε επιπλέον πυρομαχικά σε μια κατάσταση η οποία είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Μόνο μια ευρύτατη πολιτική συνεννόηση θα τερματίσει αυτή τη σύγκρουση. Κύριε Φρόιντ, λυπούμε, μόλις μου είπαν τώρα πως έχετε ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ λοιπόν, συνεχίστε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δίκιο είχα αυτή τη φορά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να σταθεί η, της, η χώρα στα πόδια της και οικονομικά μετά τους βομβαρδισμούς. Να ξεφύγει από το χάος και τον ε, πόλεμο γιατί πάλι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν είναι η Αλκάιντα και το Ισλαμικό κράτος με άμεσες συνέπειες στην Ευρώπη. Από ό,τι μας λένε ένας από αυτούς που χτύπησαν στο Παρίσι είχε εκπαιδευτεί στην Ιεμένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στο σύστημα, ζητώ συγγνώμη, δεν έφταιγα εγώ. Λοιπόν, Ιγνάσιο Κοράο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε περίπου 3.000 ε, άμαχοι πολίτες ε, και πάρα πολλοί άλλοι νομίζω ότι αρκεί για να κατανοήσουμε την κατάσταση στην Εμένη. Αυτό δεν είναι καινούριο. Η Εμένη έχει εμπλακεί σε αυτή την κατάσταση εδώ και πολύ καιρό. Πάντως ε, έχει εξελιχθεί η κατάσταση, μεγάλες δυνάμεις έχουν εμπλακεί, οι οποίες όμως μεγάλες δυνάμεις δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ότι είναι δικοί μας φίλοι. Γιατί μου φαίνεται ότι έχουν προτείνει πάρα πολλά, έχουν φτιάξει ωραία προγράμματα, ε, ειρηνευτικά λένε να παρέμβουν, αλλά δεν νομίζω ότι επικρατεί σαφήνεια στο να πούν ότι η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι η βασικά εμπλεκόμενη πλευρά, ότι δεν θα τη πουλάνε όπλα. Γιατί κατ' ουσίαν η Ιταλική κυβέρνηση είναι εκείνη που πουλάει τα όπλα ε, προσφέρει και πουλάει επίσης ε, και βόμβες ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. και εμείς είμαστε πολύ αδύναμοι στο να μπορούμε να παρακολουθούμε αυτά που μας λένε οι επικεφαλείς στην εξωτερική πολιτική. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί έναντι της Σαουδικής Αραβίας. Ο επόμενος στον κατάλογό μου είναι ο κύριος Φρανσίσκο Ασσί τον οποίο δεν βλέπω στην αίθουσα. Άρα ε, δίνω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, στην κυρία Μικέλα Γκουφρίντα, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η κατάσταση στην Ιεμένη είναι πραγματικά ολέτρια. Ε, πάνω από 80% των πολιτών χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλάμε για 21 εκατομμύρια ανθρώπους ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα κάθε μέρα και χειρότερα ε, και στα νοσοκομεία και στους χώρους υποδοχής. Βεβαίως η κατάσταση δεν είναι χειρότερη από τις άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, αλλά η Εμένη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μεμονωμένη περίπτωση εμφύλιου πολέμου. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο κατ' ουσίαν αφορά όλη την περιοχή. Η, η Εμένη είναι χρόνια ολόκληρα το πεδίο μάχης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, σύγκρουση ανάμεσα στο Ριάντ και ε, στο ε, Αμάν. Έτσι λοιπόν τα δικαιώματα των πολιτών στην Ιεμένη ε, καταπατώνται. Αυτό είναι ανησυχητικό. Πρέπει να στηρίξουμε τα Ηνωμένα Έθνη για να έχουμε άμεσα και και πάυση πυρός. Δεν πρέπει να ξεκινάμε μόνο από την ε, την αντιμετώπιση, αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του ζηλωτισμού. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, θα δώσω το λόγο και στους τρεις. Ο πρώτος είναι ο κύριος Στάνισλα Πότσακ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, εκτιμώ τις ε, προσπάθειες των ευρωπαϊκών οργάνων στην προσπάθειά τους να λύσουν την κρίση στην Ιεμένη. Δυστυχώς όμως ε, είναι κρίμα που ε, το μόνο που κάνουμε τελικά είναι να παρακολουθούμε απρακτή την σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας σε αυτή τη χώρα. Ε, έχει σημασία και το τι χρηματοδότηση δίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ντροπή, θα έλεγα, αυτό που συμβαίνει, λαμβάνοντας υπόψη το πόσο υποφέρουν οι κάτοικοι τη Ιεμένη. Ε, η Σαουδική Αραβία εδώ και καιρό προσπαθεί να γίνει εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, αλλά ο ρόλος της στην περιοχή είναι τουλάχιστον ύποπτος. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτές οι χώρες, το και η Σαουδική Αραβία, να μην φέρονται σαν η Εμένη να είναι η πίσω του αυλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιωμένη είναι τραγική. Περίπου τα τρία τέταρτα χρειάζονται βοήθεια. Ε, υπάρχει λοιπόν ο πόλεμος αυτός, μένεται ο πόλεμος, ε, ο πόλεμος ανάμεσα στην Ισαντική Αραβία και το Ιράν για να ε, κατακτήσουν την περιοχή. Η κατάσταση επιδεινώνεται τα Ηνωμένα Εθνή έχουν δώσει επίπεδο 3 στην ανθρωπιστική κρίση, το πιο υψηλό επίπεδο. 20 εκατομμύρια ανθρώπων χρειάζονται επιγόντω ανθρωπιστική βοήθεια. Οι βόμβες ε, δεν ε, φίδονται κανενό. Ε, πρέπει να δοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Τι τελευταίε ημέρε, για άλλη μια φορά, πλήγει ένα νοσοκομείο με γιατρού χωρί σύνορα θα πρέπει να βελτιωθεί η υποδομή, να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια, να μην πλήττεται ο άμαχος πληθυσμός, γιατί όλα αυτά επιδεινώνουν την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υψώσει τη φωνή της ε, για να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα προς την κατεύθυνση μιας ε, πολιτικής λύσης. Ευχαριστούμε και ελευταίος ο κύριος Νότης Μαριάς, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τον περασμένο οκτώβριο ο επικεφαλής του ερυθρού σταυρού δήλωνε ότι η ιεμένη μετά από πέντε μήνες πόλεμο μοιάζει με τη συρία μετά από πέντε χρόνια πόλεμο. από το μάρτιο του 2015 έχουν χάσει τη ζωή τους δέκα χιλιάδες άνθρωποι εκ των οποίων πολλοί άμαχοι και μεταξύ αυτών εξακόσια τριάντα παιδιά. ταυτόχρονα εκτιλήσεται μια μεγάλη κλίμακα ανθρωπιστική κρίση καθώς σύμφωνα με τον οηε από το 21 εκατομμύρια πληθυσμό τα 19 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό τα δεκατέσσερα δεν έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και περίπου τριακόσιες είκοσι παιδιά υποσιτίζονται λόγω του εναέριου και ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η σαουδική αραβία σε μια χώρα που εισάγει το 90% των αναγκών της. μετά από τον βομβαρδισμό ενός καταβλισμού προσφύγων σχολείων και μονάδων υγείας ήρθε να προσθεθεί στη λίστα των παράπλευρων απολειών χτύπημα σε ιατρικό κέντρο των γιατρών χωρίς σύνορα ενώ ταυτόχρονα η αραβική συμμαχία κατηγορείται από διεθνείς παρατηρητές ότι κάνει χρήση βομβών διασποράς. η ευρωπαϊκή ένωση έχει ηθικό καθήκον να αναγνωρίσει τα εγκλήματα πολέμου που τελούνται στην ιεμένη. η επιτροπή πρέπει να προτείνει μέτρα κατά των εθνώντων. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον τελευταίο ο κύριος για την Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο πράγματι σωστά υπογραμμίστηκε. Δεν είναι δυνατόν απλώς να παρακολουθούμε απρακτή. Δεν είμαστε απλώς παρατηρητές ε, και δεν, δεν πρέπει να είμαστε και δεν είμαστε παρατηρητές. Όλοι σας ε, είπατε ότι ανησυχείτε με την κατάσταση στην Ιεμένη. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα μέλη του Συμβουλίου και μιλώντας εξ ονόμου τη κυρίας Μογκερίνη μπορώ να πω το ίδιο. Ε, προσωπικά έχω επισκεφθεί επανειλημμένω στην Ιεμένη και η κρίση αυτή ήταν προβλεπόμενη. Ε, η διακυβέρνηση ήταν πολύ κακή επί πολλά χρόνια, ε, η προστασία του περιβάλλοντος ήταν μηδαμινή, της κληρονομιάς κλπ. Έτσι έχουμε φτάσει σε μια καταστροφική κατάσταση. Ε, όλοι οι, όλες οι οργανώσεις που χορηγούν βοήθεια την περιγράφουν με τον ίδιο τρόπο, οπότε όλοι μας ανησυχούμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα παραμείνουμε παρατηρητές ή όχι. Ε, η, ο δραστήριος ρόλος της, της εκπροσώπου είναι ε, το γεγονός ότι μπορεί να μιλήσει με όλους και η κρίση αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο αν, ε, λάβουν, αν λάβουν μέρος όλοι και μόνο αν γίνουν αλλαγές προόδου και σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό σημείο, το κλειδί της υπόθεσης. Βέβαια, υπάρχουν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ε, και εδώ βέβαια δεν μιλώ ως κυβέρνηση της Ολλανδίας. Ε, είναι σαφές όμως ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υιοθέτησε ένα συμβαστικό ψήφισμα στις 2 Οκτωβρίου 2015 που καθορίζει τους όρους για την λειτουργία μιας Εθνικής Επιτροπής Έρευνας την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ότι θα λειτουργήσει ανεξάρτητα και το υπογραμμίζω αυτό προκειμένου να διερευνήσει όλες ε, τις ε, καταγγελίες παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει στενά ε, μέσω της είπα της εκπροσώπου τις συνεδριάσεις και τα πορίσματα αυτής της Επιτροπής. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε όχι μόνο στην ανθρωπιστική κατάσταση, αλλά και τον σεβασμό στον, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Και αυτό μας ανησυχεί, γιατί ε, αναφέρεται η χρήση πυρομαχικών σε ε, κατοικημένες περιοχές. Η, ο υπάτος εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα το, το ανέλαβε, ε, ανέλαβε δράση και συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά τα όπλα. Ε, αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι ένα εμπάργκο στη Σαουδική Αραβία δεν αποτελεί απάντηση, ε, όμως ε, ε, από το 2008 υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου η οποία θα συζητηθεί ξανά στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, αναρωτιέστε για τις περιφερειακές διαστάσεις αυτού του θέματος συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και άλλων ε, χωρών της ε, περιοχής. Ε, καταρχήν, ε, δεν θα, θα πρέπει να αποφύγουμε η κρίση αυτή να διαβρινθεί. Και όλοι μας στηρίζουμε τις συνομιλίες για την Ιεμένη ε, θα πρέπει οι συνομιλίες αυτές να διατηρηθούν, να προστατευθούν και ασφαλώς να σημειωθεί πρόοδος σε επόμενες μέρες. Ελπίζουμε ότι η διαδικασία αισία θα συνεχιστεί παρόλο ότι ε, περιμένουμε καθυστερήσεις. Οι αποτελέσματα στις αρχές Φεβρουαρίου μάλλον είναι ε, δύσκολο να επιτευχθούν η ε, ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ε, έχει ταξιδέψει πάρα πολύ στην περιοχή προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία. Μας ικανοποιούν οι δηλώσεις της κυβέρνησης της ε, Ιεμένης και των αρχών της Σαουδικής Αραβίας που είναι, δείχνουν δεκτικότητα και ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστεί μια παύση πυρός που θα διαρκέσει και θα, η λύση θα βρεθεί σύμφωνα με το ψήφισμα 2260 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Και αυτό το έθιξαν πολλά μέλη του ε, Ευρωκοινοβουλίου. Ε, τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε επιθέσεις εναντίον των γιατρών του κόσμου σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτό ασφαλώς θα πρέπει να διαρευνηθεί. Και περιμένω ότι ο ύπατος εκπρόσωπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης να μας αναφέρει για αυτό το θέμα στις ε, μελλοντικές συζητήσεις τις οποίες ανέφερα. Το ερώτημα είναι φτάνουμε μέχρι την... Ε, αν ε, δίνουμε το χέρι στην Τεχεράνη, ναι, γιατί υποστηρίζει η Τεχεράνη της, την ειρήνευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει ε, τις Ιρανικές αρχές να παίξουν ένα ε, θετικό ρόλο γιατί η, το Ιράν έχει μεγάλη σημασία. Αν δεν υποστηρίξει τη διαδικασία το, το μόνο που απομένει, ε, οι μόνοι που θα βγουν κερδισμένοι είναι το Ισλαμικό κράτος και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για την Ιεμένη. Είναι επίγον το θέμα, αλλά αν δείτε και τα νούμερα ε, των ανθρώπων που βασανίζονται, γίνεται φανερό ότι το θέμα έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Η σταθερότητα στην Μέση Ανατολή, μάλλον η αστάθεια της Μέσης Ανατολής, μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια και σε μας και ανασφάλεια. Ε, η ειρήνευση ε, θα δώσει όχι μόνο πολιτική ε, δεν θα αποτελέσει μόνο πολιτικό άλμα αλλά θα βοηθήσει και στην ανακατασκευή ε, την αναδόμηση της χώρας και της πόλης ανά ιδιαίτερα. Εμείς ε, θα κινητοποιήσουμε όλους μας τους εταίρους ε, έτσι ώστε η διεθνής κοινότητα να ακολουθήσει μια συνολική σφαιρική προσέγγιση και καλούμε και τις ε, αρχές της ε, Ιεμένης ε, να παίξουν το θετικό του ρόλο. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτά τα οποία μας είπατε. Τελείωσε η συζήτηση.